Ξεκινάμε τι εργασίε, αν έχει την καλοσύνη. Σχέδιο μερίσιας διάταξης θεωρείται εγκεκριμένο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, υπάρχουν αντιρρήσει, δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Μία έχω. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πακέτο για την κινητικότητα έχει γίνει εκ νέου επίκαιρο. Ελήφθη απόφαση της ομάδας ΕΛΚ το πρωί για να μας ενημερώσει το λόγο ο κύριος Βιλ Βαντεκάμπ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είπατε ότι σήμερα το πρωί πράγματι στην ομάδα του ΕΛΚ, στην Επιτροπή Μεταφορών και χθες Κουβεντιάσαμε το θέμα, συζητήσαμε τα διαδικαστικά που αφορούν το πακέτο κινητικότητας υπαριθμών 1 εμπνευστήκαμε θετικά θα έλεγα από τις αποφάσεις των συνεδριάσεων των συντονιστών, τη συνεδριάσεως των συντονιστών που έλεγε χώρα την προηγούμενη Δευτέρα και από τις συζητήσεις που ακολούθησαν στην Επιτροπή Μεταφορών. Εμπνευστήκαμε από όλα αυτά λοιπόν και τελικά οδηγηθήκαμε σε μια νέα συζήτηση στην Επιτροπή μας ε, στο ΕΛΚ και θα από πλευράς διαδικαστικής λοιπόν Μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, αλλάζουμε θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, διαφωνούμε με το περιεχόμενο, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει ακόμα να αποφασιστεί. Ευχαριστώ, Βιμ Βαντεγκάμπ, για την ενημέρωση. Για κατανοητούς λόγους, προτιμώ μια νέα απόφαση των συντονιστών να ληφθεί και να ενημερωθεί διόντως η Επιτροπή Μεταφορών πριν στείλω επιστολή στον πρόεδρο Ταγιάννη. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή απουσιάζουν κάποιοι συντονιστέ σήμερα, θα ήθελα σήμερα να είχαμε συνεδρίαση συντονιστών μετά συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά δεν είναι όλοι εδώ. Προτείνω λοιπόν γραπτή διαδικασία με προθεσμία Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Έτσι θα ξέρω ποια θα είναι η θέση κάθε πολιτικής ομάδας και θα στείλω έτσι την επιστολή με την αναγκαία βεβαιότητα για την πλήρη ενημέρωση του Πρόεδρου Ταγιάννη και των Πρόεδρων των Ομάδα. Ε, Ηρίστον παρόδο, η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 7 Φεβρουαρίου για να είσαστε πλήρως ενημερωμένοι για τη διαδικασία, σας τα λέω αυτά. Σας προτείνω λοιπόν να ζητήσετε από τον κύριο Βίκερ γρήγορα να μας στείλει γραπτό σε ένα briefing με ενημέρωση όσον αφορά τις διαθέσιμες επιλογές σε περίπτωση που θα πάμε στην Ολομέλεια. Συμφωνείτε? Ωραία. Ο κύριος Χέρτογκ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ορίστε. Ναι, να πω κι εγώ ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι για το τι θέλετε να στείλετε, τι θα περιέχει αυτή η επιστολή, ποιο θα είναι το περιεχόμενο. Ποιος είναι ο, στόχο μας, ο στόχος μας. Αν χρειάζεται να στείλουμε αυτή την επιστολή, αν χρειάζεται να αποκτήσουμε μία πλειοψηφία. Δεν, καταλαβαίνω γιατί θέλετε να στείλετε επιστολή στον ε, πρόεδρο Ταγιάννη. κύριε Χέρτουγκ. Vous avez pu voir, il y a eu un changement de décision. Άλλαξε απόφαση. Η πρώτη επιστολή ήδη απεστάλλει. Διότι είπαμε ότι η άσκηση των Προέδρων θα έπρεπε να αποφασίσει, δεν υπήρχε πλειοψηφία στην Επιτροπή. Απεστάλλει λοιπόν η επιστολή. Ο ρόλο εμού τη Προέδρου ποιο είναι. Να βεβαιώσω ότι υπάρχει πλειοψηφία στου συντονιστέ. Γι' αυτό την Παρασκευή πριν τι 12 έχετε περιθώριο να μα πείτε αν κάποια ομάδα θα πάει στην Ολομέλη ή όχι. Από τη στιγμή που θα έχω μια πλειοψηφία θα ξαναστείλω μια επιστολή όπως Σύμφωνα με τη διαδικασία στον πρώτο Ταγιάννη να πω ότι πρέπει να μπει το θέμα στην ημέρηση διάταξη ολομέλειας. Το καταλάβατε. Ηλίου φαϊνότερον. Ο Βάλτερ θα μας εξηγήσει τη μέθοδο. Όμως ήμουν ξεκάθαρη, έτσι. Ορίστε, ορίστε. Η επιστολή που απεστάλει στον πρόεδρο δεν ευνοούσε καμία λύση. Εξηγούσε την κατάσταση και ότι δεν ελήφθη απόφαση σε επίπεδο επιτροπής. Αν αλλάξει η πλειοψηφία στην επιτροπή και έχουμε πλειοψηφία των ομάδων που θέλει να πάει στην Ολομέλεια με το θέμα, αυτό μπορεί να εκφραστεί μέσω δεύτερης επιστολής στον Πρόεδρο και να θεωρηθεί σε μια νέα θέση της Επιτροπής Τραν. Αυτή είναι η επιλογή. Γι' αυτό η κυρία Ντελή προτείνει να στείλουμε δεύτερη επιστολή, που ακολουθεί την πρώτη, πρώτερη επιστολή. Κύριε Έρτουγκ, δεν θέλω να ανοίξουμε τώρα συζήτηση. Συγγνώμη που αναλαμβάνω, λέει ο Λοιπόν, κάτι υπόθηκε. Από ό,τι κατάλαβα, να στείλουμε επιστολή, είπατε. Για να ζητήσουμε κάτι για τα διαδικαστικά. Ίσως δεν κατάλαβα καλά επειδή η πλειοψηφία στην Επιτροπή Μεταφορών είναι ξεκάθαρη, μπορείτε να στείλετε επιστολή διευκρινιστική, όπως μπορείτε να αποκαλέσω, στον πρόεδρο Ταγιάννη, αλλά όχι πλέον για το θέμα αν θα πάμε στην Ολομέλεια ή όχι. Αυτό έχει ήδη ξεκαθαριστεί ή όχι. Και πρόεδρος, μου λέτε ότι δεν είμαι καλή καθηγήτρια με άλλα λόγια. Λοιπόν, είναι σαφέστατο. Μία επιστολή απεστάλη στον κύριο Ταγιάννη, διότι δεν υπήρχε πλειοψηφία, έγινε αυτό. Είπαμε, η διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασίσει. Σήμερα υπάρχει μια νέα πλειοψηφία. Πρέπει να πω λοιπόν ότι έχετε μέχρι τι 12 την Παρασκευή να πείτε θέλουμε να πάμε στην Ολομέλεια, δεν θέλουμε να πάμε στην Ολομέλεια. Μπορώ να του πω ότι έχω πλειοψηφία θέλω να πάει στην Ολομέλεια και το λέω στην επιστολή στον κ. Ταγιάννη, Επιτροπή Μεταφορών ζητά να πάει στην Ολομέλεια. Τελεί και παύλα. Τελείωσε. Συμφωνεί. Ωραία. Ε, κύριε Κασέσκα και μετά. Προχωράμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη. Δεν έλαβε χώρα ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών. Όπου ίσως η πλειοψηφία να είχε τοποθετηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση μέσω ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφοφορία δεν έγινε. Αυτή η μορφή δράσης είναι κάπως ανεπίσημη και δεν αποτελεί βάση αυτή η σωστή για λήψη απόφασης. Αυτό είναι το, δεύτερο, το πρώτο, το δεύτερο που θέλω να θίξω. Τι ψηφίζουμε. Εάν γίνει ψηφοφορία, τι θα ψηφίσουμε και πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Αν δύο από τα τρία τμήματα του πακέτου απορριφθούν και ένα εγκριθεί, τι θα γίνει. Στείλτε μου παρακαλώ πληροφορίες. Επί ποιας βάσος αποφάσισαν οι συντονιστές ότι αυτό το πακέτο θα πρέπει να προωθηθεί. Εγώ δεν είδα επί ποιας βάσος οι συντονιστές ε, πήραν αυτή την απόφαση. Τι βάση χρησιμοποίησαν. Το πρώτο που έχω να πω Κάθε πολιτική ομάδα πρέπει να καταλάβει ότι ο ρόλος του συντονιστού είναι και ένας ρόλος εμπιστοσύνης, σας εκπροσωπεί. Αν ο κύριος Βιμ το βλέπει αυτό, εγώ δεν μπήκα στη θέση του ΕΛΚ. Πιστεύω ότι ο εκπρόσωπος, ο συντονιστής θα πρέπει να γίνεται σεβαστός στην τοποθέτησή του. Αν έχω ένα αίτημα εκ μέρους του ΕΛΚ. Δεν θα πάω στην ομάδα και να πω ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί, όχι. Δεν θα κάνω εγώ κάτι τέτοιο. Είσαστε μεγάλοι. Όταν συντονιστής παίρνει μια απόφαση και αποστέλει μια επιστολή επίσημη στην Πρόεδρο, η Πρόεδρος εισακούει το περιεχόμενο και φροντίζει του ώστε η απόφαση ε, να ληφθεί υπόψη. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικαστική συζήτηση όσον αφορά τι θα πρέπει να ψηφίσουμε μπλα μπλα κλπ. Αυτά θα τα συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε στις εργασίες μας. Δεν έχω καμία επιθυμία σήμερα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Υπήρξα σαφέστατη όσον αφορά το τι θα κάνουμε, κυρίως για το αίτημα για την Ολομέλεια. Δηλαδή, Δεύτερη επιστολή θα αποσταλεί. Πριν από αυτό οι συντονιστέ θα πρέπει να στείλουν ένα mail και να πούν ναι ου αν θέλουν να πάνε στην Ολομέλεια και μετά θα αποσταλεί επιστολή για να ζητήσουμε εν ονόμως Επιτροπής Τραν αυτό το θέμα να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Συμφωνείτε? Ο κ. Βιμ Βαντεκάμ. Και μετά κλείνω τα μικρόφωνα, γιατί εγώ θέλω να προχωρήσω. Ε, κοιτάξτε κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι διαδικαστικά μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια Μπορούμε διαδικαστικά να κινηθούμε στην Ολομέλεια. Αυτό δεν προδικάζει στο ποιο θα πάει στην Ολομέλεια και πώ θα πάνε τα πράγματα. Θέλω να αναφερθώ στη συνεδρίαση τη επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να ξέρουμε ποια πρόταση θα πάει τελικά με αυτή τη συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Και θα δούμε αν θα γίνει ψηφορία με την Τραν, χωρίς την Τραν ή επί της αρχικής προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχόλησης. Έχουν πολλά πράγματα να συμβούν που θα πρέπει όλα αυτά τα στάδια και βήματα να τα προετοιμάσουμε προσεκτικά. Κύριε Λιπεράσκη, ο τελευταίος που θα πάρει το λόγο, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην καλή βούληση των συντονιστών να αποφασίσουν τι θα γίνει. Από αυτό που καταλαβαίνω, ψήφισαν το περασμένο καλοκαίρι το θέμα, το πρόθεσαν οι συντονιστές και απεστάλει στην Επιτροπή Μεταφορών και πριν από μερικές μέρες ψηφίσαμε το θέμα, αλλάξαμε την έκθεση του κυρίου Έρτογκ σε ένα από τα τρία τμήματα, όχι στα άλλα τμήματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, η απόφαση που Ελήφθη για το θέμα τον Ιούλιο δεν ισχύει τώρα. Επαναλαμβάνω, δεν θα ξανανοίξουμε τη συζήτηση τώρα. Όσον αφορά αυτό που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, θα γίνει συνεδρίαση συντονισμού την επόμενη εβδομάδα. Θα αφορά τη μέθοδο συζήτηση και δεν θέλω να κουβεντιάσω μαζί με εσά που δεν συμφωνείτε με το συντονιστή σα, αν ο συντονιστή σα αποφάσισε σωστά ή όχι. Έχετε μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι συνεννοηθείτε. Είσαστε μεγάλοι. Δεν θα κάνω εγώ τη δική σα τη δουλειά. Αν δεν συμφωνείτε με τη θέση του συντονιστού σα, να του το εξηγήσετε και να διαπραγματευτείτε μαζί του ποια θέση πρέπει να λάβει πριν το mail που θα στείλουμε. Ωραία, ξεκάθαρα. Συνεχίζουμε με ένα θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον διότι θα ασχοληθούμε με την έκθεση Κλόντια Σμιθ, πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αφορά τις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αφορούν τη μεταφορά εμπορευμάτων. Κυρία Σμιτ, καλημέρα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα και έντονη συζήτηση, γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα και βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε μέχρι και 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η έκθεσή μου έχει πιο τεχνικό χαρακτήρα, γι' αυτό πιστεύω ότι καταφέραμε ε, τόσο σε επίπεδο πολιτικών ομάδων όσο και σε επίπεδο χωρών να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά με στενή συνεργασία. Το θέμα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί καιρό και θα έχει μεγάλες επιπτώσεις. Στην έκθεση προσπαθούμε να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη διάφορων προτύπων IT στις εμπορευματικέ μεταφορές, τα οποία θα χρησιμοποιούνται ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ενισχύσουν την οικονομία της Ένωσης. Ε, γίνεται λόγος για ψηφιοποίηση, για ε, οχήματα χωρίς οδηγό κτλ. Είναι τομείς οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν απασχολήσει και τομείς στους οποίους έχουν εντοπιστεί ελλείψεις. Ε, όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσει πόρους και ταυτόχρονα χρόνο, νομίζω είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει έτσι. Ε, τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να δημιουργήσει πρότυπα για την επικοινωνία με τις ε, αρμόδιες αρχές. Καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και έλεγχο των εμπορευματικών μεταφορών. Έτσι θα διασφαλιστεί και η ε, σωστή μεταφορά των ε, δεδομένων. Αν παρατηρήσουμε τι συμβαίνει, θα δούμε ότι στο 99% των εμπορευματικών μεταφορών ε, παρατηρούνται κάποια μικροπροβλήματα. Όμως ε, υπάρχουν ορισμένοι τομείς που θέλουν προσοχή, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η μεταβατική περίοδος που χρειάζεται για αυτές να είναι κάπως μεγαλύτερη έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ε, αγοράσουν το υλικό που χρειάζεται για την ε, ψηφιακή αυτή μετάβαση. Κατόπιν, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι είδαν την πρόταση αυτή όχι ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Ελπίζω λοιπόν στην ψηφοφορία να επιτύχουμε μια δυνατή πλειοψηφία και η έκθεση να συνεισφέρει στο επόμενο βήμα, αν όχι να λύσει το πρόβλημα. Ε, πρέπει να δεχτούμε την ηλεκτρονική λοιπόν μεταφορά των δεδομένων, αλλά και να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στις επιχειρήσεις να ε, περάσουν σε αυτό το στάδιο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι με λυπεί το γεγονός πως η έκθεση αυτή, παρότι είναι πάρα πολύ σημαντική, εξετάζεται τώρα στο τέλος τη κοινοβουλευτική θητείας. Ελπίζω η επόμενη, το επόμενο κοινοβούλιο να μάθει από τα λάθη του και να μην τα επαναλάβει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σμιτ. Θα ξεκινήσουμε την ε, συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους και για τη δουλειά που έγινε από κοινού με διάφορες προτάσεις και με ένα κοινό όραμα. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος η πρόταση είναι να δώσουμε κίνητρα όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την καινοτομία και με αυτό που είπε η συγγήτρια όσον αφορά τον όλο χρονισμό και από την άλλη πλευρά, αυτή ήταν η διαδικασία, από την άλλη πλευρά για το περιεχόμενο. Δηλαδή θέλουμε το ταχύτερο δυνατόν να καταλήξουμε σε μεταφορές χωρίς τη χρήση χαρτιού και αυτό για τη μείωση του κόστους αλλά και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων που γνωρίζουμε ότι τώρα είναι ένα κενό το οποίο δεν έχει καλυφθεί και θα διευκολύνουμε επίσης τον έλεγχο από πλευράς αρχών και ελπίζω ότι αυτή η μείωση του άχθους του διοικητικού να γίνει κάτι αισθητό το ταχύτερο δυνατό με την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και ότι οι εμπορευόμενοι ταυτόχρονα θα μπορέσουν να αρπάξουν αυτή την ευκαιρία που γεννάται από την καινοτομία αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές μεταφορών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επενδύσεις που ήδη έχουν γίνει από τους εμπορευμένους. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να ε, ποστούν ζημίες. Και δεν θα πρέπει να ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι ουδέτερα για να μην κυριαρχούν κάποιες πλατφόρμες για την αλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε συμπεριλάβει και σε άλλες εκθέσεις που συζητήσαμε σε την Επιτροπή. Γι' αυτό πιστεύω ότι ακολουθούμε σωστή κατεύθυνση και ελπίζω σύντομα το κείμενο να εγκριθεί. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Και εμεί ευχαριστούμε, κύριε Μνηματέ. Κύριε Ζε... και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σμιτ. Επίσης και τους κύριους εισηγητές γιατί καταλήξαμε σε μια πολύ καλή έκθεση, την οποία μπορούμε να υποστηρίξουμε. Σε κάθε περίπτωση, αν μπορούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, αυτό είναι καλό και πρέπει να γίνει. Είναι προφανές ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι πιο ε, απλά και πιο εύκολο να χρησιμοποιούνται από ότι τα έντυπα. Υποστηρίζουμε λοιπόν την εκθέση Σμιτ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε κυρία Λοτόφσκη. Κυρία Μπιλμπάου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. να συγχαρώ και εγώ την κυρία Σμιτ για το έργο της και επίσης για τους, ε, να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες για τη βοήθεια. Καταλήξαμε σε συμβαστικές λύσεις, με συζήτηση και πιστεύω ότι ο βασικός στόχος αυτής της έκθεσης που εντάσσεται και στο πακέτο για την κινητικότητα είναι να διευκολυνθεί η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσουμε προς μια ε, κατάσταση περισσότερης ψηφιοποίησης και με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Διαπιστώνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακαιρματισμό στην αγορά, ότι έχουμε πολλά διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα που δεν ε, λειτουργούν, δεν, δεν είναι διαλειτουργικά, δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις ε, αρχές. Πιστεύω ότι με τι συμβιβαστικέ λύσει τι οποίε καταλήξαμε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι διαλειτουργικό, και αυτό θα βοηθήσει και τα κράτη-μέλη και τις ιδιωτικές εταιρείες έτσι ώστε εφαρμόζοντας αυτό το νέο σύστημα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και να γίνουμε ως Ευρώπη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να αποκτήσουμε μια ηγετική θέση και με αυτόν τον τρόπο επίσης να φροντίσουμε έτσι ώστε η μεταφορά των εμπορευμάτων να ρηπαίνει λιγότερο, να είναι πιο αποτελεσματική για το περιβάλλον. Μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση έτσι ώστε αυτή, αυτά τα μέτρα να αρχίσουν να εφαρμόζονται από την επόμενη θητεία. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Καλώς ήρθατε κυρία... Έχετε το λόγο. Υποστηρίζουμε και εμείς την έκθεση Σμιτ, πιστεύουμε ότι πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Χαιρόμαστε επίσης για το γεγονό ότι ακολούθησε και από τις προτάσεις μας. ε, οι οποίε πήγαιναν προ κατεύθυνση να επισημάνουν ότι όταν έχουμε ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο ήδη λειτουργεί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε. Ε, είναι σωστό αυτό και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις μικρές ε, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι η συγγήτρια δεν ακολούθησε όλες τις προτάσεις μας που είχαν ε, περισσότερο σχέση με το περιβάλλον. Ε, και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Για τα θέματα αυτά θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πιο μακριά στον τομέα των μεταφορών. Θα θέλαμε να είχε δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές τις προτάσεις, δηλαδή στην κλιματική αλλαγή. Γνωρίζουμε ότι οι μεταφορές είναι ο μόνος τομέας της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου αυξάνονται οι εκπομπές. γνωρίζουμε ότι έχουμε δεσμεύσει για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, τι οποίε πρέπει να ακολουθήσουμε και θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι πιο αποτελεσματικέ λύσει σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε, κύριο Πακά. Παχά. Ζητώ συγγνώμη, δεν θέλατε να πάρετε το λόγο. Κυρία Κόζευσκάι, είστε καλύτερα με το, το, το γόνατο που έχετε χτυπήσει, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Κυρία Πρόεδρε, τη συνάδελφοι, θα είμαι σύντομη αυτή τη φορά. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω και να, τις, ε, και να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές, καθώς επίσης και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Γιατί στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ψηφιοποίηση, απλοποίηση και μεγαλύτερη χρήση των λύσεων πληροφορικής στον τομέα των μεταφορών. Θα υποστηρίξουμε τις συμβαστικές τροπολογίες πιστεύουμε ότι βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση προς την πρόταση της Επιτροπής. Προσπαθούμε δηλαδή να γίνει ο κανόνας η χρήση των ηλεκτρονικών εντύπων στον τομέα αυτόν. Και θα ήθελα να επενθυμίσω και στους ορισμένου συναδέλφους που πήραν το λόγο ότι χρειαζόμαστε ένα εναρμονισμένο και νομικά δεσμευτικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και για τις ε, ε, ε, εταιρείε τι μεταφορικέ και για όλες τις εταιρείε στην Ευρώπη. Όπως έλεγα λοιπόν, υποστηρίζουμε και την έκθεση και τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Έχω μια διευκρινιστική ερώτηση, την οποία κάπως μου απάντησε και η συγγήτρια. Λέμε ότι από τη μια θα πρέπει εν τέλει να, δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιούν όλοι οι, όλες οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον, στο χώρο. Γιατί, γιατί χρειαζόμαστε ένα πλήρας και ε, σύστημα το οποίο ε, μόνο έτσι θα διασφαλίσει ότι τα έντυπα είναι, οι πληροφορίες ανταλλάσσονται με τρόπο τυποποιημένο. Απ' την άλλη όμως πρέπει να προβλέψουμε και μία μεταβατική περίοδο, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην αναγκαστούν ξαφνικά να χρησιμοποιούν τις ε, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πριν η αγορά μάλιστα να δημιουργήσει διαφορετικές ανταγωνιστικές πλατφόρμες για να μπορέσουν να επιλέξουν μία από αυτές. Επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και να το αναλύσουμε σε μεγαλύτερο βάθος κατά πόσον μπορούμε με τον κανονισμό να φροντίσουμε, να προσπαθήσουμε να ε, εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα και σε περιπτώσεις διεθνών μεταφορών που καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις. Δεδομένου ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις διεθνείς συμβάσεις, θα πρέπει να το αναλύσουμε σε μεγαλύτερο ε, βάθος για να μην υπάρξει ανασφάλεια δικαίου ή οποιοδήποτε πρόβλημα ε, σε σχέση με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Το έργο της ήταν εξαιρετικό επί του θέματος αυτού. Και είμαι βέβαιη ότι μπορεί το σύνολο της Επιτροπής μας να υποστηρίξει ε, το αποτέλεσμα. Αυτά. Ευχαριστώ. Και εμείς. Ευχαριστούμε. Κυρία Σμιτ. Έχετε το λόγο ω συγγήτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια, τα παραδικά σα λόγια, τα οποία με βοήθησαν. Δυστυχώς έχουμε μείνει αρκετά πίσω και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα σωστά μέτρα και να κάνει τα κατάλληλα βήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σμιτ. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Θυμάστε τις κάρτε σα. Να ελέγξουμε πρώτα απ' όλα αν υπάρχει απαρτία. Είμαι σίγουρη, αλλά α ελέγξουμε. Ψηφοφορία δοκιμαστική. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένα λεπτάκι, θα ψηφίσω κι εγώ, λέει η πρόεδρος. Υπέροχα. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη συμβιβαστική 7, υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 50. Θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει. Ελέγχουμε για την τροπολογία 55. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Αδίκιο έχετε. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε για την 57. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. με μικρή διαφορά απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 10 εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ομού δύο τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πάμε τώρα στο 98 και το 100 μαζί υπέρ κατά αποχές Δεν είναι ξεκάθαρο. Κάποιοι έχουν κουραστεί και δεν σηκώνουν τα χέρια τους. Λοιπόν, ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφορίας. Και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τι έγινε εδώ. Δεν σηκώνετε το χέρι σας. Δεν φταίνε τα μάτια μου. Δεν φταίει η πρόεδρος. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Α, κατά αυτή Ε, 99. Ε, ωραία. Συμβαστική 15 λοιπόν. Υπέρ κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, 34 μάλλον υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Το σύνολο λοιπόν του κειμένου όπως τροποποιήθηκε το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Et le Πέρας ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Σμιτ, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεσή σας. Et nous continuons Συνεχίζουμε πρόταση του κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληροφορίες τις σχετικές με τις εμπορευματικές μεταφορές. Μία ψήφα έχουμε. Ηλεκτρονικός πώς θα λάβει χώρα. Oui, oui, c'est le règlement 11. Et c'est pas le transport des marchandises Non, c'est ce qu'on vient de voter. Ah, oui. Nous votons le rapport de Madame Desmonté. Στην έκθεση Δελμόντε, όσον αφορά τους κανόνες και τις κοινέ προδιαγραφές που αφορούν τους οργανισμούς που μπορούν να πραγματοποιούν επιθεώρησης επισκέψεως των λιμένων σε περίπτωση αποσύρσεως του Ηνωμένου Βασιλείου θα τροποποιηθεί ο κανονισμός 391-209. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clos. 35 υπέρ. Με μεγάλη διαφορά υιοθετείται. Συγχαρητήρια κυρία Τερμόντε. συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της καταξιδοδότησης συμπράξεως όσον αφορά τις προδιαγραφές των συστημάτων, εφιών, συνεργασίμων συστημάτων μεταφορών. Η κυρία Γκάσιν Μάισνερ είναι η συγκεκριά. Έχετε το λόγο. Περιμένετε κυρία Μάισνερ. Α, μου λένε ότι πρέπει να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Ποιο. Α, δεν έφτασε ακόμα εκπρόσωπο της Κομισιόν. Θα περιμένουμε να αποχωρήσουν οι αποχωρούντες glaube, jetzt kann es losgehen, oder? Μπορώ τώρα να ξεκινήσω. Ehrlich gesagt, ich weiß, was die Kommission... Ε, για να είμαι ειλικρινής, ξέρω τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εντάξει, ας περιμένουμε πρώτα να μιλήσει, να κρατήσουμε την ε, σειρά. Είμαι εισηγήτρια, πολύ σωστά, όμως εδώ πρόκειται να ακούσουμε την ε, παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα πρώτα θα μιλήσουν εκείνοι και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σχολιάσει. Ναι, το ξέρω ότι εσείς θα μιλήσετε πρώτοι. Είναι έτοιμη η Κομισιόν. Ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μάισνερ, διότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν έχει καταθέσει ακόμα. Κατέφτασε, είναι εκεί. Ποιο θα μιλήσει εν όνομα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Ορίστε, έχετε το λόγο. Μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ το απόγευμα. Διότι μπορούμε τελικά να πούμε ότι το μέτρο που ετοίμαζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ευφύ μεταφορικά συστήματα δημοσιεύτηκε στην θερίδα για την καλύτερη νομοθεσία, στην πύλη για την καλύτερη νομοθεσία και είναι πολύ καλό βήμα. Μα στηρίξατε επανειλημμένα εσεί. Αναγνωρίζοντα τη δυνατότητα που έχουν τα ευφύ συστήματα μεταφορών για την οδική ασφάλεια αλλά και για την αποτελεσματικότητα τη κυκλοφορία και διευκολύνεται και αυτόματη κινητικότητα και μα δίνει την ευκαιρία, την ευκαιρία στην Ευρώπη να προηγηθεί αυτή η σημαντική εξελίξεω. Από παθητική ασφάλεια περάσαμε σε ενεργητική ασφάλεια και τώρα σε συνεργαστική ασφάλεια. Το 2019 έγινε το σημαντικό βήμα. Εντοπίσαμε όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Ξεκίνησε καλά ο χρόνο. Δημοσιευθήκαμε στην πύλη μα το θέμα για την καλύτερη νομοθεσία και το τελικό μέτρο ε, για 15 Μαρτίου ελπίζουμε να το υποβάλουμε. Να υπενθυμίσω εντάχει περί τίνο επρόκειτο για τον καταξιδότηση κανονισμό να μιλήσω. Στόχος, ασφάλεια δικαίου και ευρύ εφαρμογή του συστήματος. Περιμέναμε, περιμέναμε επί μακρόν για αυτά τα συστήματα. Καλύπτουμε συνεννόηση οχήματος με οχήματα και όχημα με υποδομή. Βασικός στόχος είναι η διαλειτουργικότητα, η συμβατότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχονται. Για να επιτευχθεί αυτό αντιμετωπίζουμε τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο, ασφάλεια. Αν θέλουμε κάθε χρήστη του δρόμου, κάθε όχημα και κάθε υποδομή, κάθε στοιχείο να συνομιλούν μεταξύ του, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Οι υπηρεσίε πραγματικά. Τι μηνύματα θα πρέπει να ανταλλάσσονται. Πρέπει να είναι εύληπτα σε όλη την Ευρώπη τα μηνύματα. Και κατανοητά. Τρίτον, το δυσχερέστερο, η τεχνολογία αν όλοι πρέπει να συνδέονται, δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να το συζητήσουμε αυτό. Τώρα, είναι σημαντικό να τονίσουμε κάτι. Αυτός ο κατεξοδότηση κανονισμός είναι η βάση, είναι το πρώτο βήμα και πολλά ακολουθούν. Εντοπίσαμε αρχικό κατάλογο υπηρεσιών και αρχικό τρόπο χρήσεως αυτών και αναπτύξεως αυτών. Πολλές ε, αλλαγές αναμένονται, πολλές υπηρεσίες θα προσθεθούν συμπληρωματικές τεχνολογίες θα αναπτυχθούν και θα προσθεθούν. Το όφελος από την υφιστάμενη κάλυψη Φερρυπίν. Η κατεξοδότηση πράξη έχει κάλυψη όσον αφορά το μέλλον, είναι μελλοντοστραφής, αλλά θα πρέπει να είμαστε και συμβατοί με τη βάση. Αυτό είναι βασικό στοιχείο. Διότι εφ' αυτού δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια, να δώσουμε ασφάλεια σε αυτούς που χρησιμοποιούν το σύστημα σήμερα. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι συνδέονται σήμερα θα παραμείνουν συνδεδεμένοι και δεν θα έχουμε έτσι συνέχεια των υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά να πω ότι είμαι ευχαριστημένο που είμαι εδώ, διότι είμαστε στην τελική ευθεία του σημαντικού αυτού έργου και των εξελίξεων που έχουν κρατήσει μια δεκαετία τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βάντερ Λίντεν, για αυτή τη λακωνικότατη παρουσίαση. Έχουμε όμως πολλές ερωτήσεις. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εντάξει, τώρα είναι η σειρά μου. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς όταν γίνεται λόγος για FEE, e, συστήματα μεταφορών και συνδεδεμένα οχήματα, να προσέξουμε πάρα πολύ για να δούμε τι είναι πραγματικά αναγκαίο έτσι ώστε να συνοδεύσουμε την πρόοδο με τα κατάλληλα μέτρα. Ε, φυσικά, ε, να πω ότι με ευχαριστεί πολύ το ότι αναφερθήκατε στην εμπιστοσύνη και στην προστασία δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση αυτή την θα, θα πρέπει να προσέξουμε να προασπίζουν ακριβώς ε, την προστασία αυτή. Νομίζω πως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς διότι μπορεί να σημειωθεί τεράστια πρόοδος Για φανταστείτε τώρα τα, αυτο, τα οχήματα να μπορούν να επικοινωνήσουν. Αυτό, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα βοηθήσει πάρα πολύ τις ε, μεταφορές και την οδική ασφάλεια καθώς και την ομαλή διεξαγωγή της ε, κυκλοφορίας. Φυσικά αυτό δεν γίνεται χωρίς προστασία των δεδομένων, γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρατε. Δεν έχω τίποτα να πω εναντίον της παρουσίασής σας, νομίζω πως φαίνεται ότι το έχετε σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Είναι απέραντες οι δυνατότητες που έχουμε στο μέλλον και μάλιστα ο άντρας της κόρης μου ασχολείται με τον ε, τομέα αυτόν και πραγματικά είναι ένα τομέα με μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι γνωρίζω σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Ο κύριος Βιμ Βαντενκόμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά πράξεις κατά εξουσιοδότηση και γιατί αυτό έχει γίνει αντικείμενο τόση οδρυμίας κριτικής. Οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, έχω δεχτεί μεγάλη πίεση από διάφορες ομάδες και αυτές οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση έχουν δημιουργήσει αρκετές ανησυχίες. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση κυρία Πρόεδρε, είναι ποια είναι η δική μας θέση. Φυσικά γνωρίζω πως έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση για τις πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση και συνεχίζονται αυτές οι διαβουλεύσεις μέχρι το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τελειώνει ο χρόνος. Θα διακόψουμε για τις ευρωεκλογέ σύντομα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι επιτρέπεται να πούμε και τι όχι. Εντάξει, είμαι ευγενικό άνθρωπο, όμω θέλω να ξέρω και τα δικαιώματά μου. Δεύτερη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη φορά. Η ουδετερότητα της τεχνολογίας τι ρόλο παίζει διότι μου φαίνεται πως οι αποφάσεις έχουν ληφθεί κάπως μονόπλευρα, όπως για παράδειγμα για τα σύρματα δίκτυα, για το Wi-Fi και πως δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι τεχνολογίες. Ήδη έχουμε περάσει στη χρήση τεχνολογίας 5G και χρησιμοποιούμε τεχνολογία εχμής στην ε, κινητή τηλεφωνία. Ε, υπάρχει λοιπόν μια μεταβατική διάταξη στο σημείο 3 όπου αναφέρεται ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσθεθούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έχετε κάνει αυτό. εξελίξεις ε, λαμβάνουν χώρα ταχύτατα. Η τεχνολογία αλλάζει από στιγμή σε στιγμή. Όμως ε, αυτό το τεχνολογικά ουδέτερη νομίζω πως ε, δεν θα βοηθήσει τη διαλειτουργικότητα. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν εκπροσωπούνται εξίσου στην πρόταση της Επιτροπής. Θεωρώ λοιπόν πως δεν δίνουμε στις νέες τεχνολογίες τη θέση που τους αρμόζει. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της. Επίσης, ε, αυτόνομη οδήγηση. Έχω δει από πρώτο χέρι τις εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη όλες ε, τις ε, διαφορετικές πτυχές των τεχνολογικών εξελίξεων. Επίσης, έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν τις ε, συνδέσεις ανάμεσα στα θέματα αυτά, αλλά η απάντηση της Κομισιόν παραμένει ασαφής. Υπάρχει συμβατότητα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και της πράξης κατεξουδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίμαντα Κάμπ για να απαντήσει στα ερωτήματά σας διότι θέσατε ένα άμεσο ερώτημα. Να γνωρίζετε την ώρα έχουμε λάβει το σχέδιο της κατεξοδότησης πράξεως, αλλά όχι την τελική κατεξοδότηση πράξη. Αυτό ήταν ένα σχόλιο που αφορούσε και το ερώτημα σας. Κύριε Έρτουγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και εγώ έχω μια ερώτηση παρόμοια με εκείνη του κυρίου Βάντεκαμπ. Θα ήθελα να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται στο ε, κομμάτι της ε, τεχνολογίας και ποια είναι τα στοιχεία που σας οδήγησαν υπέρ της μίας μορφής τεχνολογίας, του Wi-Fi ας πούμε, αυτό που αυτή τη στιγμή αν βλέπω καλά, επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 5G από την άλλη. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Wi-Fi που λείπουν από το 5G και αντίστροφα. Αυτό λοιπόν θα ήθελα ε, να μου το απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχω μια άλλη ερώτηση για όλους και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν θέλουμε να εδραιώσουμε την τεχνολογική ουδετερότητα στις πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση, θα πρέπει να προσέξουμε την ε, διατύπωση. Όμως, χρειάζεται να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή, μπορούμε να λάβουμε μια τέτοια πολιτική απόφαση σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Έτσι, το λέω για να το πω. Θα με ενδιέφερε λοιπόν όμως να μάθω όντως αυτές τις διαφορές ανάμεσα στις δύο μορφές τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κίλονεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτηση η δικιά μου είναι πολύ παρόμοια με αυτές των συναδέλφων προς την Επιτροπή γιατί πιστεύω ότι η πρόταση που μας έρχεται για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση δεν είναι τεχνολογικά ουδέτερη. Ενώ έχουμε πολλές φορές μιλήσει υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητας, το θέμα το έχει αναδείξει ως πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και από την Επιτροπή. Επίσης, εγώ δεν έχω καθόλου πιστεί για, την... για το κατά πόσο θα υπάρχει ασφάλεια δικαίωση σε ολόκληρη την Ευρώπη όταν δεν ορίζουμε την έννοια της τεχνολογικής, ε, τη γνώμη της διαλειτουργικότητας. Και παρόλα αυτά το χρησιμοποιούμε ως λέξη καθημερινά. Βεβαίως δεν πρέπει κανείς να ποντάρει μόνο σε μια τεχνολογία. Αυτό έχει κινδύνους. Ήδη είναι, ε, αμφισβητείται το κατά πόσον το 5G είναι το κατάλληλο πρωτόκολλο για, για δίκτυα ITS όταν έχουμε μεγάλες ροές κυκλοφορίας. Εάν επίσης και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες οι χρήστες που στην πραγματικότητα θα πληρώσουν για αυτές. Οι πεζοί, επίσης οι ποδηλάτες και τι θα χρειάζεται να γίνει για να διατηρηθούν οι διάφορες τεχνολογίες και στο, επίπεδο που πρέπει. Ελπίζω να προβληματιστεί για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μόνο που υπάρχει σήμερα στο draft είναι μια φράση που λέει ότι θα μπορέσουμε να προσθέσουμε και κάποια τεχνολογία στο μέλλον. Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού ή fair play μεταξύ των ε, διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν επιλέγουμε τελικά μια συγκεκριμένη επιλογή, πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί. Γιατί υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με αυτούς που την προωθούν γιατί κατά την άποψή μου θα έπρεπε όλοι να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε, αυτή την... σε αυτόν τον ανταγωνισμό, σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ κυρία Κίλωνεν. Ε, και εγώ σκιώδης, λέει η πρόεδρος, θα ήθελα να πάρω το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση, αλλά έχω πολλές ερωτήσεις. Πρώτον, πήκυνται οι ευρωεκλογές πλησιάζουν γρήγορα. Και έχετε θέσει μια προθεσμία, σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Βάντεν Κάμπ, που είναι η 15η Μαρτίου. Λοιπόν, δυστυχώς, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει επί της ουσίας τα υπέρ και τα κατά ε, για αυτό το, πάνω σε ένα τέτοιο κείμενο, αναρωτιέμαι, μπορεί να μας εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το κείμενο θα το έχουμε εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορέσει να ασκήσει και το καθήκον του και τα δικαιώματά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβόλιο. Γιατί αυτό που έχουμε λάβει αυτή τη στιγμή δεν είναι το τελικό κείμενο και για να είμαι ειλικρινής δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι στις 15 Μαρτίου θα είναι όλοι οι συνάδελφοι παρόντες εδώ. Το είπε και η κυρία Κινούνε και θα το επαναλάβω είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της προστασίας των, ε, προσωπικών ε, δεδομένων. Είναι κρίσιμη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και βλέπω στην αιτιολογική σκέψη 29 αναφέρεστε στην θετική γνώμη του ε, επόπτη προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Αρχής. Έχετε λάβει τέτοια γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα προσωπικά δεδομένα, γιατί εμείς πάντως δεν έχουμε λάβει κάποιο κείμενο σχετικό. Και ο κύριος Βαντερκάμ και ο κύριος Χέρτοκ αναφέρθηκαν σε ένα θέμα που είναι σημαντικό για μας. Ακούμε όλους να μιλούν για τεχνολογική ουδετερότητα. Και μας προτείνει τώρα μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση η οποία προωθεί μια συγκεκριμένη τεχνολογία έναντι άλλων. Ε, το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρο γιατί εσείς η Επιτροπή και όχι εμείς ο συνομοθέτης να αποφασίζει, από πού και ως πού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποφασίζει, δεν έχει και ο συνομοθέτης, ο συνομοθέτης είναι εκείνος που έχει δικαίωμα να λάβει τέτοια απόφαση. Πολύ απλή ερώτηση. Μετά. Μας λέτε ότι αυτά τα συστήματα δεν θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του 2019. Και ε, τότε γιατί βιαζόμαστε όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χώρο μας λένε ότι δεν θα είναι έτοιμοι. Μετά, θα συμφωνήσω με τον κύριο Βάντερ Κάμπ, που λέτε ότι υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες, το ανέφερε και η κυρία Μάισνερ, η τεχνολογία 5G. Ε, Λέω λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι θα προστεθεί και η τεχνολογία 5G στην ε, πράξη κατ' εξουσιοδότηση, εξυπνοείται ότι θα πρέπει να είναι συμβατή με την προηγούμενη, με τις τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται. Ε, τότε σας ρωτώ, τι εννοείται διαλειτουργικότητα. Γιατί εν τέλει ο νεοαφιχθής, η νεοαφιχθής σαν νέα τεχνολογία να πρέπει να είναι συμβατή με την προηγούμενη και όχι το αντίστροφο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα δημιουργήσει πάρα πολύ ε, δεν θα γίνει πολύ ακριβό μάλλον να αναπτυχθεί αυτή η νέα τεχνολογία. Επίση, λέτε ότι θα δημιουργηθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα είναι σε θέση να εξετάσει κατά πόσο είναι όριμη η τεχνολογία. Ποιο θα την ορίσει αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Έχω βαρεθεί τι ομάδε εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξηγήστε μου ποιο θα επιλέξει τη σύνθεση αυτή τη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Που θα, και με ποια κριτήρια αυτοί οι εμπειρογνώμονε θα αποφασίσουν αν μια τεχνολογία είναι όρημη ή όχι. Θα είστε εσεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εμείς που έχουμε και κάποια διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας μας. Επίσης, εάν είναι τα κράτη-μέλη εκείνα που πιέζουν για να, προωθηθεί αυτή, να προωθηθούν αυτές οι εκτελεστικές πράξεις, βλέπετε ότι ταυτόχρονα προβληματιζόμαστε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προσπάθησα, προσπάθησα με τρόπο ξεκαθαρό να πω ότι θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η δημοκρατία. Σας ευχαριστώ κύριε δικέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλά ερωτηματικά ακούστηκαν, δεν εκπλήσωμαι. Και έχω τρία σχόλια πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια κατεξουσιοδότηση πράξη για, για ποσόστοση σαρδελών στο, στη Νότια Ευρώπη. Εδώ είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια εν γέννη και για την βιομηχανία και την οδική ασφάλεια. Καταφθάνει υπό τη μορφή κατεξοδότηση πράξεως. Δεν ξέρω αν διαβάσατε τις 223 σελίδες των τεχνικών λεπτομεριών. Το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο τεχνικά. Λοιπόν, έχουμε κατεξοδότηση πράξη. Και δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά του το Κοινοβούλιο. Ενδεχόμενη ένσταση κατά της ε, κατεξοδότησης πράξης, πώς δρομολογείται. Χρόνια συζητάμε το θέμα. Πώς τελικά καταλήγουμε σε κατεξοδότηση πράξη για πρόταση όπου δεν μπορούμε εμείς να τοποθετηθούμε επί της κατεξοδότησης πράξεως. Με εκπλήσει αυτό. Δεν ξέρω πώς θα περάσει αυτό. Ε, και είναι πολύ σημαντικό το θέμα για να υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Πέρα το διαδικαστικό και τη μορφή. Το ανέφερα κάποιοι συνάδελφοι. Η επιλογή που γίνεται μου δημιουργεί προβληματισμό. Γιατί γίνεται αυτή η επιλογή όταν κάπου όπως τις είπα δεν έχει γίνει κάποια επιλογή ή άλλη επιλογή όπως στην Κίνα που είναι οι μεγάλοι παίκτες στο παγκόσμιο προσκήνιο. Θα μπορούσαμε ίσως να μην αποφασίσουμε αμέσως. Καμία τεχνολογική ουδετερότητα και συμβατότητα Ανοδική, καθοδική, δεν είμαι ειδικό. Αλλά νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα. Τεχνολογικά προβλήματα και επενδυτικά προβλήματα. Δεν έχω την κατάλληλη εκπαίδευση. Δεν κατανοώ τα τεχνολογικά επιχειρήματα. Τα παραρτήματα είναι κάπως αποθαρρυντικά. Μήπως Χρειάζεται πολιτική συζήτηση πρώτα το θέμα. Ουδετερότητα τεχνική να είναι υποχρεωτική. Προστασία δεδομένων. Αυτά είναι κυρίως πολιτικά θέματα. Μήπως αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και να είναι πιο εύληπτη συζήτηση και μήπως αυτή η κατεξοδότηση πράξη δεν είναι ιδανική μορφή αντιμετωπίσεως του θέματος. Ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για να ε, προβάλλει ένσταση. Όχι ότι είναι εναντίον. Πρέπει να σταματήσει αυτή η διαδικασία όπω ξεκίνησε. Αυτή η προσέγγιση με ανησυχεί ο τρόπο αντιμετώπιση του θέματο και η διαδικασία με προβληματισμό. Μην ανησυχείτε, κύριε Ρικέ, λέει πρόεδρο. Ελέγχουμε το θέμα, το ελέγχουμε. Θα ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Βαντερλάντεν, έχετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα προσπαθήσω να απαντήσω διαδοχικά σε αυτά που υπόθηκαν. Αρκετοί ομιλητέ Αναφέρθηκα στην προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Πράγματι είναι βασικά στοιχεία. Στοιχεία που πρέπει να συζητηθούν, αλλά δεν μπορούν να αποφευχθούν. Στόχος της προσπαθία μα είναι η βελτίωση της ασφάλειας και η βελτίωση της κυκλοφορία. Πώ μέσω τη διαβίβαση στοιχείων. Από την αρχή που υπάρχει διαβίβαση στοιχείων, η προστασία των δεδομένων γίνεται θέμα. Δεν μπορεί να αποφευχθεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε το εξή. Αυτό ο κατεξισοδότηση κανονισμό δεν δίνει οριστική απάντηση στην αντιμετώπιση του προβλήματο. Ο κατεξοδότηση κανονισμό λέει σαφώ ότι πράγματι ο κανονισμό, ο γενικό προστασία δεδομένων ισχύει πλήρω. Αυτό είναι το πλαίσιο που έχουμε στην Ευρώπη για τη μετώπιση των θεμάτων προστασία δεδομένων. Η κατεξοδότηση πράξη τι κάνει. Σαν ένα τμήμα του κεφαλαίου ασφαλείας παρέχει πολλά στοιχεία για ελαχιστοποίηση των ανησυχιών για την προστασία των δεδομένων. Επί παραδείγματι, κάθε μήνυμα που τα μελλοντικά οχήματα θα ανταλλάσσουν είναι ανώνυμο. Και αυτή η ανωνυμία αλλάζει συνεχώς. Έτσι δεν περαιτέρω τα συστήματα θα μοιράζονται μόνο τα στοιχεία που είναι απόλυτα αναγκαία ούτω ώστε να παρέχει την υπηρεσία. Τέλο, εξαρτάται από εκείνου που αναπτύσσουν την τεχνολογία, χρησιμοποιούν τεχνολογία και τι υπηρεσίες παρέχουν και επιλέγουν να εξασφαλίσουν αυτοί ότι συμμορφώνονται πλήρω με τον κανονισμό, το γενικό ύπνος των δεδομένων. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εντό του κατεξοδότηση αυτού κανονισμού, λέει ο μιλητή. Δεύτερον, Κάτι που προσέχθηκε όλος ιδιαίτερο, σχεδόν όλοι οι ομιλητές το έθεσαν. Το θέμα της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας. Τι γίνεται με τις μελλοντικέ τεχνολογίες. Καταρχάς, να ξεκινήσω από κάπου. Ρωτήσατε τι προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει αλλαγή ρυθμού, να πετύχει αλλαγή ρυθμού όσον αφορά ε, την οδική ασφάλεια. Να τη βελτιώσει δραστικά. Και γι' αυτό θέλουμε να συνδέσουμε όλους τους χρήστε των δρόμων για να το κάνουμε αυτό πρέπει να συζητήσουμε τεχνολογία. Πώς θα διασυνδεθούν όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου. Απλούστατα σήμερα αυτό που βλέπει κανείς τον κανονισμό αυτό είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή σήμερα. Δεν είχαμε εναλλακτική. Ελπίζαμε μάλιστα ότι αυτή η εκδοχή του κατεξιδότηση κανονισμού ήδη θα εμπειρήχε δύο εναλλακτικέ. Αν θυμόσαστε αυτό που γράψαμε το 2016 Ρητά είχαμε πει ότι αυτό που χρειαζόμαστε στον τομέα είναι η βρυδική προσέγγιση στην ε, τεχνολογία επικοινωνιών. Τι εννοούσαμε με αυτό. Συμπληρωματικές τεχνολογίες. Διαφορετικά ωφέλη για διαφορετικές υπηρεσίες. Ελπίζαμε να έχουμε τουλάχιστον δύο από τις συμπληρωματικές τεχνολογίες ήδη να υπάρχουν σήμερα. Δυστυχώς αυτό ήταν ανέφικτο διότι δεν έχει οριμάσει ακόμα η εφαρμογή των τεχνολογιών. Θα γίνει, είμαστε πεπισμένοι. Γι' αυτό είπα στην πρώτη μου παρέμβαση, πολλές αλλαγές και τροπολογίες αναμένονται. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που προτείνουμε σήμερα πράγματι είναι διαλειτουργικό. Τι σημαίνει αυτό. Εξασφαλίζουμε ότι αν κάποιο από εσά, οποιοδήποτε από σας πάρει το αυτοκίνητό του ή τη μοτοσυκλέτα του ή φορτηγάκι ένα βαρύ όχημα ένα πούλμαν, αν το οδηγήσει στην Ευρώπη αυτό το όχημα και συναντήσει οποιοδήποτε άλλο όχημα, ότι τα οχήματα θα συνεννοηθούν, θα καταλάβουν το ένα το άλλο. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό σημαίνει για μας η διαλειτουργικότητα. Και με τα θλίψεις μου λέγω ότι απαιτεί πολλές τεχνικές λεπτομέρειες στα παρατήματα. Κατανοώ πλήρω ότι είναι περίπλοκο το θέμα, ε, δυσνόητο αλλά η ουσία δεν είναι τόσο δύσκολη. Η ουσία είναι ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι κατανοούν ο ένας τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Μια άλλη ερώτηση που ετέθη. Τι ρόλο παίζουν οι μελλοντικές τεχνολογίες, πώς συμπεριλαμβάνονται Πρέπει να θυμηθούμε και σημαντικό ότι αυτό που συμπεριλαμβάνουμε στον κανονισμό είναι εφαρμόσιμο μόνο για αυτέ τι πρώτε υπηρεσίε, αυτή την ομάδα υπηρεσιών, τι πρώτε υπηρεσίε που παρέχονται. Με άλλα λόγια, αν μελλοντικέ τεχνολογίε καταφτάσουν, που θα καταφτάσουν, το ξέρουμε, τι αναμένουμε ότι θα δώσουν νέε υπηρεσίε. Υπηρεσίε που θα χρειάζονται, θα απαιτήσουν νέε τεχνολογίε. Αυτό δεν δημιουργήσει πρόβλημα με τον παρόντα κανονισμό. Αυτό που λέγουμε είναι ότι αν κάποιος τα σημερινά μέσα τα χρησιμοποιήσει, θέλουμε να ωφεληθούν αυτές τις υπηρεσίες αύριο επίση. Με τη... Η τεχνολογία, κυρίως στην πληροφορική, εξελίσσεται τάχιστα. Δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια όμως για τα οχήματά μας. Αν αγοράσει κανείς ένα αυτοκίνητο σήμερα, θέλει να δουλεύει και αύριο και σε 10 χρόνια. Γιατί η μέση ηλικία ενός οχήματο είναι 15 χρόνια ο κύκλος ζωής του. Αυτό που δεν θέλουμε είναι αυτά τα οχήματα σε δύο χρόνια να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες υπηρεσίες. Κυρίως επειδή γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσουμε τα συστήματα ένα σημαντικό τμήμα του στόλου πρέπει να έχει εξοπλιστεί των οχημάτων. Αυτό χρειάζεται χρόνο. Και πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε τα δέοντα. Με άλλα λόγια, αν ρωτήσετε ποιε εναλλακτικέ έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε και μέχρι να ολοκληρωθεί το 5G και αν ήταν καλή ιδέα να αναπτύξουμε το 5G, θα είχαμε τη συζήτηση και θα λέγανε κάποιοι. Μισό, μισό λεπτό, είναι σχεδόν έτοιμο το 6G, θα είναι καλύτερο. Ας περιμένουμε για το 6G. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Κύριε Βίμαν Δεγκάπ. Eh, Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε το συντομότερο αυτές τις πράξεις κατά Δεν πρέπει να χρονοτριβούμε. Θα ήταν ανόητο. Γιατί όμως να επιλέξουμε μια τεχνολογία η οποία ήδη ε, υφίσταται αρκετές πιέσει. Η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα και θα έπρεπε οι πράξη κατά εξουσιοδότηση να μας δίνουν το περιθώριο να μπορούμε να αναπτύσσουμε γρήγορα τις νέες τεχνολογίες. Στον φάκελο για την αυτόνομη οδήγηση δεν γίνεται λόγος για το Wi-Fi ή για την ε, κινητή ε, τεχνολογία, το ζητούμενο είναι να βγουν τα οχήματα στο δρόμο. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο ότι ο, η πράξη αυτή καταξιοδότηση προβλέπει μία μόνο μορφή τεχνολογίας. Η Επιτροπή Μεταφορών θα συζητήσει ξανά το θέμα αυτό για την αρμοδιότητά μας, αλλά όπως είπε και ο Ισμαήλ Ερτούγκ είναι επίγοντα θέματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει γιατί έχει κάνει αυτές τις επιλογές. Το ζητούμενο είναι να, να χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες γρήγορα. Η κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Να παρατήρησα πως ήμουν μάλλον θετική σε σχέση με τους συναδέλφους μου. Όμως ε, αυτή η θετική μου στάση ίσως οφείλεται στο ότι έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και στην ε, ιδιωτική μου ζωή. Μπορώ να συμφωνήσω και εγώ με τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νέα αυτή τεχνολογία θα είναι επαναστατική, θα οδηγήσει σε περισσότερη οδική ασφάλεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντική είναι και η προστασία των προσωπικών δεδομένων και όπως σας είπα ε, προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και με την τεχνολογική ουδετερότητα. Όπως ε, είπατε κι εσείς, έχουμε τώρα Wi-Fi, τώρα 5G, 6G, θα λίγο θα έχουμε και 7G κατά πάσα πιθανότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια. Και εμείς πρέπει να συνοδεύσουμε την ε, τεχνολογία με τα μέτρα που θα βοηθήσουν σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με αυτό που υπάρχει σήμερα στο εμπόριο. Και για μένα είναι φυσικά κατανοητό και αυτονόητο. Σίγουρα ασχολούμαστε πάρα πολύ καιρό με το, τα θέματα αυτά. Όμως ε, πρέπει να δράσουμε τώρα. Η 15η Μαρτίου δεν είναι νωρίς. Το αντίθετο. Χρειάζεται να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, διότι βαδίζουμε προς μια κατεύθυνση άγνωστη. Και σίγουρα υπάρχουν φόβοι, το ακούσαμε. Τι γίνεται με την ε, ασφάλεια των πεζών σε περίπτωση αυτόνομης οδήγησης οχημάτων χωρίς οδηγό. Φυσικά και υπάρχει φόβος ε, για λάθη. Δεν χρειάζεται λοιπόν ε, μόνο διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία σίγουρα δεν πρέπει να πηγαίνουν σε λάθος χέρια αλλά και προσοχή στην ε, εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Και σίγουρα το άγνωστο τρομάζει. Το καταλαβαίνω αυτό. Ε, σας ξαναλέω, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα αυτό και δεν έχω τόσες πολλές ερωτήσεις όσο οι συνάδελφοι γιατί το έχω ψάξει. Αλλά θεωρώ σωστό την επιλογή της πράξης κατά εξουσιοδότηση, διότι θα ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις εξελίξεις. Και αυτή η προσαρμογή για μένα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για μια τεχνολογία άγνωστη δεν μπορεί να λάβει από τώρα αποφάσεις για το, μέλος, ε, για το μέλλον. Πρέπει να συνοδεύσουμε τις εξελίξεις. Τώρα δεν έχει σημασία το τι κάνουν οι Κινέζοι, τι κάνει ο ένας ο άλλος. Το θέμα είναι στην Ευρώπη να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα και να διασφαλίσουμε αυτήν την διαλειτουργικότητα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάισνερ. Ωστόσο πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπροστά μας το τελικό κείμενο της πράξης. Επομένως δεν γνωρίζουμε ακριβώ πότε θα μας το αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το draft, το προσχέδιο. Και δεν είναι... δεν γνωρίζουμε ποιο ακριβώ, θα είναι το τελικό κείμενο. Δεύτερο, είναι το ζήτημα των προθεσμιών, του χρονοδιαγράμματος. Λυπάμαι, αλλά φοβάμαι ότι θα έρθει πολύ καθυστερημένα το τελικό κείμενο. Και δεν υπάρχει ο χρόνος για να γίνει η συζήτηση με τρόπο δημοκρατικό και με διαφάνεια όπως πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα το θέσω ίσως το ζήτημα στους συντονιστές, γιατί νομίζω ότι επί του θέματος αυτού ίσως να χρειάζεται ένα ψήφισμα με το οποίο να εκφράζεται η θέση της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Μπορεί να αλλάζει η τεχνολογία γρήγορα, αλλά εμείς παραμένουμε συνομοθέτες. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι. Να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τις τεχνικές πυροδιαγραφές, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο συστήματα, ανάμεσα σε αυτές τις δύο τεχνικές επιλογές. Θα ήθελα να ξέρω λίγες περισσότερες πληροφορίες να έχω για να καταλάβω γιατί επιλέγει αυτό που επιλέγει η Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Χαρτοκ. Θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να μας στείλει γραπτό την απάντησή της για να μπορούμε όλοι να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Εξέφρασε λοιπόν το αίτημά μας, το σημειώνει και η γραμματεία. Θέλουμε μια γραπτή ε, απάντηση. Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Κύριε, Χερτούγκ. Ε, έλεγα λοιπόν, ε, κύριε Χέρτου για να το ακούσετε και την μετάφραση, ότι ζητήσα γραπτό να μα αποστείλει την απάντησή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι ξεκάθαρη και να την έχουμε όλοι. Εντάξει. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάλι για ζήτημα ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Καλώς ήρθατε κύριε Μαρινέσκου. Θα ακούσουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα drones, τα οποία είναι η προσγενική χρήση. Καλώς ήρθατε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την πράξη κατά εξουσιοδότηση και μετά θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κύριο Μαρινέσκου, τον εισηγητή μας. Κύριε ε, Κανέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, εξωτερικό μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε για την πρόσκληση να ε, συζητήσουμε μαζί το πολύ σημαντικό ζήτημα των ντρόουν και την πράξη κατά εξουσιοδότηση που ετοιμάζουμε για την λεγόμενη ανοιχτή κατηγορία, όπως είπατε είναι ένα προσχέδιο πράξης κατεξουσιοδότησης το οποίο ε, υποβάλαμε προς δημόσια διαβούλευση τέλος του 2018 και, και προτιθέμεθα να το εγκρίνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλη Φεβρουαρίου και μετά φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει το δικαίωμα της εξέτασης όπως πάντα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την προσέγγιση που υιοθετούμε με αυτό το προσχέδιο ε, ενός νομοθετικού πλαισίου για τα μη επανδρομένα αεροπλά, σκάφη, αεροσκάφη. Και βέβαια η πράξη κατεξοδότηση για τα drones είναι ένα, μία από τις πτυχές αυτού του πακέτου. Χρειάζεται να ε, λάβουμε μέτρα τα οποία να εφαρμόζονται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσουμε ότι η χρήση των ντρόν θα γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, ασφαλή και που θα σέβεται την ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα. Θα γνωρίζετε ότι έχει από το Σεπτέμβριο του 2018 υιοθετηθεί από την ΕΑΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις ε, ε, ε, Αεροπορικές Μεταφορές, ένας νέος βασικός κανονισμός για την ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους, και στη συνεργασία με την ΕΑΣΑ έχουμε προετοιμάσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο προσχέδια με συγκεκριμένους ε, κανόνες που θα εφαρμόζονται σε όλα τα ντρόν. Ο πρώτος θα ε, καλύπτει την χρήση των ντρόν ως οχήματα και ο δεύτερος κανονισμός θα αναφέρεται σε οποιαδήποτε άλλη χρήση των ντρόν, καθώς επίσης και τις προδιαγραφές για τις οργανώσεις τις, οποίες, τις οργανισμούς που τις χρησιμοποιούν καθώς επίσης και κάποια ελάχιστα πρότυπα για την εκπαίδευση των χειριστών τους αυτές τις προτάσεις θα τις, παρουσιάσουμε, θα τις δημοσιοποιήσουμε και θα τις παρουσιάσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, θα πρέπει να τις δούμε όλες αυτές τις προτάσεις ως πακέτο, παρά το γεγονό ότι ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες. Όμως χρειάζεται να τις δούμε ως πακέτο για να έχουμε μια πλήρη αίσθηση του τι επιδιώκει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη ρύθμιση των χώρων των ντρόων, που είναι δύσκολη αυτή η ρύθμιση, γιατί μιλούμε για μια νέα τεχνολογία η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα. Σε γενικέ γραμμέ, στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών θεωρείται ότι τα drone δημιουργούν προβλήματα, ε, αλλά αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε εκείνους που ασχολούνται με τι αεροπορικές μεταφορές. Έχουμε ανησυχίες σε σχέση με το ε, περιβάλλον, σε σχέση με τις εκπομπές τους, σε σχέση με το θόρυβο που προκαλούν ή επίσης την πιθανή χρήση τους ε, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα. Ωστόσο, τα ντρόουν, όπως οποιαδήποτε σημαντική καινοτομία τεχνολογική, μπορεί να ε, ε, δώσει μεγάλα πλεονεκτήματα στον γενικό πληθυσμό. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουμε κανονισμούς που να καλύπτουν ταυτόχρονα ένα drone το οποίο μπορεί να φτάνει τα 500 γραμμάρια μέχρι και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος το οποίο να έχει το μέγεθος και το βάρος ενός Airbus. Επομένως, πολύ διαφορετικά ε, πράγματα μεταξύ τους. Ε, Επίση, είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι ε, από startup νεοφύ επιχειρήσει στον τομέα τη τεχνολογία μέχρι αερολέσχε ή μεγάλε αεροπορικέ εταιρείε. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε μία προσέγγιση που να βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Είναι μια νέα προσέγγιση που ακολουθεί πλέον και η ΆΣΑ η ρύθμιση του χώρου των drones μας έδωσε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε αυτή τη νέα προσέγγιση. Ξεκινούμε λοιπόν από τις βασικές απαιτήσεις που η προτείνει η ΆΣΑ για, ε, και όχι τι απαιτήσει οι οποίε ήδη προβλέπονται για τη χρήση των ντρόουν ω όχημα στην νομοθεσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Επιτροπή ε, Τραν, ε, την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνεισέφερε στην υιοθέτηση του κανονισμού από την ε, πλευρά τη άσα την προηγούμενη χρονιά, αλλά επίση συνεχίσατε να συνεργάζεστε μαζί μα. Αυτό μα βοήθησε να ασχοληθούμε με ζητήματα σημαντικά όπως ζητήματα του αξιόπλου, της ε, χρήσης του των drones από αερολέσχε και του ζητήματο της ιδιωτικότητα. Με τους νέους κανονισμούς, οι αερολέσχε και τα μέλη τους θα συνεχίσουν να, μπορέσουν, να μπορούν να χρησιμοποιούν τα drone με βάση το σύστημα των αεροπορικών ε, μετακινήσεων και που, που ήδη λειτουργεί επιτυχώς μέχρι σήμερα. Οποιοδήποτε χειριστή θα πρέπει να καταγράφεται σε ένα μητρό. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εκείνου που ε, ε, χειρίζονται drone με βάρο μικρότερο των 50 γραμμαρίων, εφόσον αυτέ φέρουν κάποιον καταγραφέα που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να ε, επηρεάσει την ιδιωτικότητα. Δημιουργούμε λοιπόν ξεκάθαρες ε, διαδικασίες για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και αυτός ο αντίστοιχος κανονισμός έχει δημοσιοποιηθεί για δημόσια διαβούλευση, είναι διαθέσιμος και, και σε εσά, στα μέλη του Κοινοβουλίου. Επίσης προετοιμάζουμε ε, κατ' κανονισμό που ε, θέτει τις προδιαγραφές, τους σχεδιαστικές για τα drone που θα ανήκουν στην πλέον ευρεία και απλή κατηγορία, την ανοιχτή κατηγορία αυτές, αυτά τα ντρόν δηλαδή που θεωρητικά θα πρέπει να ε, ε, έχουν το μικρότερο κίνδυνο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει δύο, χρόνο, δύο, δύο μήνε ε, στη διάθεσή του για να εξετάσει αυτό τον ε, κανονισμό μετά την υιοθέτησή του από την Επιτροπή, όπω σα είπα, τέλη Φεβρουαρίου. Τα άλλα ντρόν, τα οποία δεν, θα καλύπτονται από αυτόν τον, τον κανονισμό, θα καλύπτονται από διαφορετική νομοθεσία. Ακολουθούμε λοιπόν μια προσέγγιση που έχει τρεις ξεκάθαρες κατηγορίες για τα μη επανδρομένα. Το πρώτο είναι η ανοιχτή κατηγορία, η λεγόμενη drone, για τα οποία δεν χρειάζεται προηγούμενη εξουσιοδότηση και οι οποίε δεν δημιουργούν μεγάλου κινδύνου. Αυτή η ανοιχτή κατηγορία περιορίζεται σε drone τα οποία δεν ξεπερνούν τα 25 χιλιόγραμμα σε βάρο και πάντοτε θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί κανεί σε ασφαλή ε, απόσταση από, από τους άλλους ανθρώπους και ε, θα πρέπει να υπάρχει άμεση διαρκής οπτική επαφή του χειριστή με τον drone του. για κάθε μια από αυτές τις κλάσεις, από αυτές τις ε, ομάδες drone ε, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές βάρους και άλλες τεχνικές προδιαγραφές και μόνο ένα drone το οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές θα μπορεί να ε, πωλείται στην αγορά. Θα πρέπει να εντάσσεται σε κάποια υποκατηγορία α1, α2 ή α3, μιλώντας πάντα για την ανοιχτή κατηγορία, το πράσινο, και ο χειριστή θα πρέπει να πληρεί από τη δικιά του πλευρά των προποθέσεων. Μετά έχουμε την ε, κίτρινη κατηγορία, την ε, υψηλότερου κινδύνου. Εδώ θα χρειάζεται μια εξουσιοδότηση, η οποία είτε θα βασίζεται σε μια αξιολόγηση κινδύνου συγκεκριμένη, για μια συγκεκριμένη χρήση, από ε, μια εξουσιοδότηση κινδύνου, κινδύνου την οποία θα κάνουν οι αρχέ, ή μια άδεια η οποία θα προβλέπει τη χρήση του ντρόν σε ένα συγκεκριμένο σενάριο, το οποίο θα περιγράφεται στην άδεια και από εκεί και πέρα θα έχουμε τους, χειριστε, ε, τους χειριστές εκείνους οι οποίοι θα έχουν πιστοποιητικό χειριστή μη επανδρομένο αεροσκάφους, το οποίο παρέχουν ήδη οι αρμόδιες αρχές. Η τρίτη κατηγορία, η κόκκινη, εδώ ε, χρειάζεται ε, εξουσιοδότηση, αδειοδότηση μάλλον, θα έχει πλοδιαγραφές αντίστοιχες με εκείνες που έχουμε για την αεροναυσιπλοεία με πιλότους σήμερα. Δηλαδή χρειάζεται ε, πιστοποίηση και του, του, φορέα που χειρίζεται, που, στον οποίο ανήκει του drone και του χειριστή. Εδώ μιλούμε για χρήση drones για την μεταφορά επικινδύνων αγαθών, για τρόουν τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν πάνω από μια συνάθρηση. Ε, οποιοδήποτε δηλαδή τέτοια χρήση η οποία θα πρέπει να περιγράφεται ε, επακριβώς και να πληρεί κάποιες προγραφές πιστοποίησης. Στην διαφάνεια αυτή βλέπετε πώς καθορίζουμε στο, στην ε, κατεξουσιοδότητα πράξη την χρήση της λιγόμενης ανοιχτής κατηγορίας, δηλαδή τους περιορισμούς που ισχύουν σε αυτήν κατά την συγκεκριμένη κατηγορία. Στην πράξη κατά ακολουθούμε επίσης και την προσέγγιση της χρήσης του σήματος CE. Αντίστοιχη προσέγγιση έχει και η άσα. Δηλαδή, θέτουμε κάποια όρια στο υψόμετρο μέχρι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιούνται, κάποιου περιορισμού απόσταση από κατοικημένε περιοχέ, την απέτηση να υπάρχει αγομεσιοπτική επαφή με το χειριστή, καθώ επίση και τον καθορισμό ορισμένων γεωγραφικών περιοχών στι οποίε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ντρο. Με όλου αυτού του περιορισμού ε, μειώνεται το, ο κίνδυνο και ε, αντίστοιχο τρόπο αντιμετώπιση του κινδύνου έχουμε δει και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, στις Ηνωμένε Πολιτείες, στον Καναδά, ε, το, η αντίστοιχη κατηγορία είναι η λεγόμενη 1-7. Ε, και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά έχουν ακολουθήσει μια ε, προσέγγιση που ανάλογα με την κλάση στην οποία εντάσσεται το drone υπάρχουν αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Όπως σας έλεγα, θα αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάσετε η ΆΣΑ και τις οποίες θα πρέπει να τις δείτε ως πακέτο. Εκεί θα θέσουμε πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ε, χρήση τους ως οχήματα, την, ε, τις άδειες που θα πρέπει να έχουν οι χειριστές και επίσης ε, προδιαγραφές τεχνικές για το αξιόπλο τους. Και όπως σας έλεγα, για τις, τα βαρύτερα ντρόν που ξεπερνούν τα 150 κιλά. Θα υπάρξουν επίσης κάποιες σχετικές προτάσεις για να αλλάξουν οι σχετικές ε, η σχετική νομοθεσία για την αεροναυσιπλοεία, για την, ε, τους ελεγκτές κυκλοφορία κυκλοφορίας, για τις γνώσεις που θα πρέπει να έχουν οι πιλότοι. Αυτά που συνέβησαν πρόσφατα στα αεροδρόμια κοντά στο Λονδίνο, Κλείσμα του Gatwick, νομίζω δείχνει πόσο σημαντικό είναι να λάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, κάποιες πρωτοβουλίε για να υιοθετήσουμε κανόνες. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Και πιστεύουμε ότι αυτές οι νέες προτάσεις που κάνουμε θα βελτιώσει τον έλεγχο που χρειάζεται να υπάρχει στη χρήση των drone. Θα πρέπει να βελτιωθεί η χρήση άμεσης ε, ταυτοποίησης ε, ε, ε, μακρισμένες ταυτοποίηση των, των drone, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστούν οι κανόνες geolocation, δηλαδή τη απαγόρευση χρήσης drone σε συγκεκριμένη περιοχή. Κάτι τέτοιο θα είχε αποτρέψει τα προβλήματα που είδαμε στο Gatwick και σε άλλα αεροδρόμια. Θα είχαν τη δυνατότητα οι αρχέ επιβολέ του νόμου να βρουν ποιο είναι αυτό που έχει παραβιάσει την νομοθεσία. Δεν ε, μίλησα για την χρήση drone για άλλες χρήσεις θα επανέλθω. Πάντως ήθελα να σας ενημερώσω, έχουμε ξεκινήσει να εξετάζουμε και άλλους τομείς. Τέλος, θα προσπαθήσουμε τα drone να είναι όσο δυνατόν πιο φιλικά προς το περιβάλλον και όσο το δυνατόν με μικρότερες εκπομπές θορύβου. Μιλούμε για ένα νέο είδο αεροπλάνου αυτή τη στιγμή, ενό ε, αερίου μέσου και θα πρέπει να φροντίσουμε οι κανονισμοί και το νομοθετικό πλαίσιο να ε, είναι ξεκάθαρο από την αρχή. σα. ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι στη διάθεσή σα να απαντήσω στις ερωτήσει σα είτε τότε, τώρα είτε τι επόμενε εβδομάδε όταν θα υιοθετήσουμε και τις της πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κορνέλη. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό των drones. Ακόμα και αν τα έχουμε καλύψει κάπως μέσω των ρυθμίσεων για την ΕΑΣΑ. Μιλάμε τώρα για κατεξουσιοδότηση πράξη. Κύριε Μαρινέσκου, θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω καταρχάς πως ε, χαίρομαι που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελευταίο περιστατικό στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειάζονται κανόνες γραπτοί κανόνες τέτοιοι που να καταφέρουν να αποτρέπεται ως το δυνατόν ε, περισσότερο τέτοια περιστατικά. Οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση λοιπόν. Ο βασικός κανονισμός ζητά στις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση να συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές ε, για την επάνδρωση, τη συντήρηση κλπ. ενό αεροσκάφους τόσο για πορική όσο και για προσωπική χρήση αλλά και για τους ε, πιλότους του αλλά και όλα τα σχετικά στοιχεία που θα διασφαλίσουν την συμμόρφωση με τις αναγκαίες προϋποθέσεις που αναφέρει το άρθρο 55. Να σας υπενθυμίσω ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται στο παράρτημα 2, το αξιόπλο, και ε, το παράρτημα 5 στους ε, πιλότους και την ε, αεροπλοία. Δεν έγινε σεβαστό το Κοινοβούλιο ε, στην ενημέρωση για αυτό το θέμα. Εκεί αναφέρεται ότι ε, δεν χρειάζεται να ε, διαβάζονται πληροφορίες για όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα, η πρόταση αυτή που λάβαμε, τι συμπεριλαμβάνει. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογής είναι μόνο για την ανοιχτή κατηγορία επιχειρήσεων. Μόνο. Δηλαδή, για drones μέχρι 25 κιλά δεν θα χρειάζεται ε, πιστοποίηση. Η πράξη κατά εξουσιοδότηση θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει ε, προϋποθέσεις ε, για τις περιπτώσεις που χρειάζονται πιστοποίηση και όχι για αυτές που δεν χρειάζεται. Δεν έχω καταλάβει εδώ τι συμβαίνει. Και τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κανονισμός. Τώρα, τα drones της ανοιχτής κατηγορίας χρειάζονται μόνο μία αξιολόγηση συμμόρφωσης και μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβεβαιώνει τις, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ε, που αναγράφονται στο παράρτημα. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ η πράξη καταξιζότητα δότηση να σταλεί και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ, διότι το 90% της πρότασης αφορά κανόνες ε, για την ε, νέα αγορά. Δεν ξέρω ακριβώ τι κάνει η Επιτροπή ΙΝΤΑ, όμως αυτά που διαβάζω ε, από την πρόταση της DigiGrow είναι αρμοδιότητα της ΙΝΤΑ. Υπάρχουν γενικές προδιαγραφές για τα drones και επίσης όπως αναγράφεται στον Γενικό Κανονισμό και όχι εδώ, υπάρχουν πληροφορίες για τον εξοπλισμό που πρέπει να εγκατασταθεί για να διασφαλιστούν αυτές οι, αυτές οι λειτουργίες. Καλύτερα λοιπόν να κοιτάξουμε και τις δύο αυτές προτάσεις, και τις ε, εκτελεστικές πράξεις και τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Αν δούμε με προσοχή λοιπόν θα ε, παρατηρήσουμε ότι γίνεται λόγος για πιστοποίηση drones. Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό και εμείς έχουμε ζητήσει πράξεις κατά εξουσιοδότηση παντού. Τώρα όμως τι γίνεται. Οι διατάξεις για την ε, πιστοποίηση των drones συμπεριλαμβάνονται στις, ε, στις εκτελεστικές πράξεις οι οποίες θα έπρεπε να αναφέρουν μόνο την ε, περίπτωση προσωπικής χρήσης και την ε, καταχώρηση ενός drone. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, η εκτελεστική πράξη αυτή ξεπερνά τις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής. Και κάτι άλλο αν θυμάστε καλά, είχατε προεδρεύσει στις ε, σχετικά με αυτό και τα 150 γραμμάρια είναι ε, πολύ σημαντικό θέμα. Στο τέλος, δεχτήκαμε να γίνει τροποποίηση στα 8 τζάουλ. Και τώρα άλλαξε το βάρος και πήγε στα 250 γραμμάρια, αλλά για τα τζάουλ τίποτα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ούτε εδώ τι έχει συμβεί. Εφόσον μάλιστα μιλάμε για ένα κείμενο το οποίο έχει τροποποιηθεί ελάχιστα. Ε, εδώ λοιπόν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ε, που θεσπίζει ο βασικός κανονισμός για την ε, καταχώρηση και οι πράξεις εξουσιοδότηση έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. τι απαιτήσει δηλαδή ως προς τον εξοπλισμό και δεν υπάρχουν διατάξεις για τις περιπτώσεις όπου ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος χρειάζεται πιστοποίηση για να μην μιλήσω ούτε για το σχεδιασμό, τον κατασκευαστή και όλες αυτές τις ε, λεπτομέρειες. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Πρέπει να το σκεφτούμε καλά πριν συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο και με πράξη κατοξιοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκου. Να δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Φώστερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιον εκπρόσωπο της ΆΣΑ που βλέπω εδώ. Φίλιπ Κορνέλης, βοήθησε αυτή η παρουσίαση που έκανες. Ήταν αρκετά ξεκάθαρη και εύληπτη. Ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μας στείλετε την παρουσίαση. Μπορείτε. Αυτό ίσως να βοηθήσει. Πριν ξεκινήσω, να σχολιάσω αυτά που συνέβησαν στο Γκάτουικ. Ούσα Βρετανοί και Λονδίνων δεν πέρασα παρατηρήτο. Ήτανε μεγάλη φασαρία. Δεν συνέβη μόνο στο Γκάτουικ αυτό. Περιμέναμε πολύ καιρό για να τοποθετηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε έναν κανονισμό και κατευθυντήριες γραμμές. Όμως στην υπηρεσία πολιτικής ε, αεροπορίας στην Ολλανδία και στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην, ε, στην Αμερική είπα είχαν κανόνες που είχαν θεσπιστεί προκαιρού. Αλλά δυστυχώς πάντα υπάρχει κάποιος ανόητος που θέλει να παίξει παιχνιδάκι ανεξαρτήτως κανόνων. Γι' αυτό εξετάσαμε και το θέμα πώς να περιφράξουμε κάποιες ζώνες, ε, κάποιες τεχνολογικές λύσεις αποκλεισμού περιοχών. Χρειάζεται σωστό σχεδιασμός συστήματα ανάγκης και οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια να κάνουν τα δέοντα. Σωστή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε άσα. Ως εισηγήτρια για την έκθεση για τα drones που υποστηρίχθηκε από την παρούσα επιτροπή, και περισσότερα από 700 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και που δημοσιεύτηκε σε επίσημη εφημερίδα το κείμενο το 2015, ε, είχαμε σαφή θέση τότε. Τι θέλαμε να κάνουμε. Αυτό θέλαμε στην έκθεσή μου. Ευπρόσδεκτη προσέγγιση. αυτό θέλαμε. Και αφορούσε και την ασφαλή χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών η έκθεση. Χρειάστηκε χρόνος έπρεπε να επανεξετάσουμε το βασικό κανονισμό. Πέρασε πολλή χρόνος από το 2015 μέχρι τώρα για να φτάσουμε σε αυτή τη θέση. Επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε. Εκεί αρχίζω να διαχωρίζω τη θέση μου από αυτή του κυρίου Μαρινέσκου. Πιστεύω ότι καλή είναι η προσέγγιση. Τότε δεν θέλαμε καν να θέσουμε όρια βάρους. Είναι γεγονός όμως ότι τα 250 γραμμάρια και κάποια άλλα κριτήρια ε, είναι η σωστή κατεύθυνση λόγω διαφόρων ειδών και τεχνολογικής προόδου και ρυθμού τεχνολογικής παρεόδου ε, μπορεί ε, σε μια εβδομάδα να γίνει πολύ πιο ελαφρύ το όχημα, να έχει το μισό βάρος και διπλάσια ταχύτητα. Ευπρόσδεκτο το σήμα CEE e της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχει συμμαχία για τα drones στο Ηνωμένο Βασίλειο που συζητά το θέμα επί μακρόν. Μίλησα και με τη Βασιλική ε, Αερολέσχη. Ε, συζητούν το θέμα. Είναι τεράστιο θέμα για όλες τις χώρες. Από τον κατασκευαστή μέχρι του τελικού χρήστη. Συμφωνούν με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρω... το CE. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Χρειαζόμαστε κριτήρια σε όλη την Ευρώπη. και εθνικές υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας πρέπει να ενημερωθούν. Αυτές έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να κάνουν τα δέοντα. Αυτά έχω να πω. Δεν είναι εύκολα αυτά τα θέματα, είναι αρκετά περίπλοκα. Καλή θέση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή άλλωστε είναι και η θέση της ομάδας μου, του ECR. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ο κ. Βαντεμπέργκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομο. Πολλά ήδη υπόθηκαν από την κυρία Φώστερ. Ευπρόσδεκτο το σχέδιο εφαρμοστική και κατεξοδότηση πράξη. Δεν καλύπτονται τα πάντα. Το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συγκεκριμένη κατηγορία βάσει προσεγγίσεως μέσω κινδύνου χρειάζονται πολλά να καλυφθούν, τα διάφορα ενδεχόμενα αυτό θέλουμε όμω, αυτή την κατεύθυνση ακολουθήσουμε. Λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση Φώστερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο κειμένου έλαβε υπόψη και συζητήσει για 250 γραμμάρια και τα κιλο Στο παράτημα δεύτερο τμήμα αναφέρονται αυτά. Πρέπει να βρούμε όμως τη σωστή ισορροπία και να μην παρέμβουμε με υπερβολική νομοθεσία στα παιχνίδια όπως αποκαλούνται, γι' αυτό έχουμε και ανοιχτή κατηγορία. Με το CE0, όπου δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσει όπως για τα μεγαλύτερα μη επανδρομένα οχήματα, αλλά η χρήση του drone και ο συγκεκριμένος κίνδυνος που είναι η συνέπεια χρήσης αυτού, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά. Έχουμε βρει σωστή ισορροπία στο σχέδιο κατεξοδότηση πράξεως, κατεξοδότηση πράξεω και τη εφαρμοστική πράξεω. Δεν πρέπει να υποβάλουμε ένσταση και να έχουμε αντιρρήσει και να χάσουμε άλλο ένα χρόνο, αλλά να τα εφαρμόσουμε αυτά. Να υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Η άσα, η βιομηχανία, οι εθνικοί εμπειρογνώμονε, όλοι συμφωνούν. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Χρειάζεται επιτάχυνση η προσπάθειά μα. Πάντα θα υπάρχουν ερωτηματικά. Και έγαχα ερωτηματικά μετά από αυτά που συνέβησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά χαίρομαι από τις εξηγήσει που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο non-paper που βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Εκεί καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν απαιτήσει σχετίζονται με γεωευαισθητοποίηση, ε, εντοπισμό των σκαφών από μακριά. Ελήφθησαν υπόψη αρκετές ανησυχίες που ακούστηκαν στους τελευταίους μήνες, ε, τελευταία χρόνια. Εγώ θα έλεγα γρήγορα να εγκριθεί η κατεξουσιοδότηση πράξη θα δώσει ασφάλεια δικαίου και στη βιομηχανία για να μπορεί να κινηθεί επί στις βάσεις και, και για τις δυνάμεις επιβολής του νόμου στα διάφορα κράτη-μέλη και τις εθνικές υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, θα βοηθήσουμε έτσι, αλλά βέβαια εξίσου σημαντικό και την ΕΑΣΑ. Ας επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ας ολοκληρωθεί το θέμα. Και ας εφαρμοστεί στην πράξη και ας λειτουργήσει στην πράξη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαν Λίντεμπουργκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Να επενθυμίσω όμως ότι υπήρξαμε σαφέστατοι με τον κύριο Μαρινέσκου μέχρι τις 6 ώρα το πρωί όσον αφορά το κείμενο της ΕΑΖΑ. Θυμόσαστε. Θέλαμε να δούμε σε ποια πράγματα ανήκουν σε εκτελεστικές πράξεις και στις εξουδότηση πράξεις και βλέποντας το κείμενο Αγνώ αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη αυτά που είπαμε τότε, τις διαπραγματεύσεις που είχαμε τότε, διότι έχω πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν και πετυχημένα στοιχεία στην πράξη. Παραδείγματο χάρη, χαίρομαι που ένα ντρόν των 250 γραμμαρίων, ένα μικρό, μη επανδρομένο όχημα 250 γραμμαρίων, παιχνίδι ντρόν, να πλαισιώνεται σωστά, με συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια. Όταν έχουμε μικρά drones, υπάρχει καταγραφή του drone και έχει αστική ευθύνη ο πιλότος. Δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικά προστατευτικοί. Θέλουμε να αποφύγουμε όμως τα τυχήματα και να προστατεύσουμε τη ζωή, την ιδιωτικότητα επίσης των ανθρώπων. Τι με εκπλήσει όμως, που υπάρχουν κάποια εκπληκτικά πράγματα σε αυτή την πράξη και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα. Π.χ. drones μέχρι 25 χιλιόγραμμα, 25 κιλά μπορούν να ύπτανται στην κατηγορία open δεν με πείθετε ότι ένα, ένα drone των 25 κιλών δεν χρειάζεται επιστοποίηση και δεν θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο πτήσης στις ελεγκτικές αρχές. Αν αύριο αρχίζουμε να έχουμε 25 κιλά drones χωρίς σχέδιο πτήσης, ποιες αρχές είναι αρμόδιες κλπ. Σας διαβεβαιώνω ότι θα γίνει χαμός. Και από την αρχή των συζητήσεων στην έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου την έκθεση της ΕΑΖΑ κατηγοριοποίησαμε τα drones και χαρακτηριστικά επικίνδυνότητα των drones. Ενέργεια, κινητική ενέργεια που θα μπορούσε να απελευθερωθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν ήταν το αγαπημένο μου θέμα, αλλά περί αυτού επρόκειτο. Αν έχουμε τα ενεργειακά κριτήρια Κομισιόν, εξηγήστε μου πώς μπορούμε να δώσουμε κανόνες στα ελαφρά ε, οχήματα και τις να μην δίνουμε κανόνες σε αυτές οι πτάμενες βόμβες των 25 κιλών. Δεν θα μπορούμε, μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει με αυτά τα drones. Γι' αυτό όταν βλέπω τις εικόνες αυτές που δείξατε, μας δείτε τρία είδη drones έχουμε. Έχουμε μία κατεξοδότηση πράξη για το ένα και τα άλλα δεν πλαισιώνονται. Οι άλλες κατηγορίες Εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Αυτές ήταν οι σκέψει μου, η μικρή μου συνεισφορά στη συζήτηση. Η κυρία Γιούζο έχει το λόγο. Θέλετε να μιλήσετε για τα drones. Κύριε Βίμ Κάμπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο Γνωρίζουμε πόσο δεινό διαπραγματευτής είναι ο κύριο Μαρινέσκου. Συχνά όμω έχει δίκιο, όταν πρόκειται για, ιδίως για νομικά κείμενα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ της βασικής νομοθετική πράξης, της, εκτελεστική πράξη εκτελεστικής πράξης και της πράξης του Δεν γίνεται αυτό. Εάν στην εκτελεστική πράξη υιοθετούμε διατυπώσεις ή όρους οι οποίοι διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της βασική νομοθετική πράξη, αυτό δεν επιτρέπεται. Εδώ ξεπερνάει τι αρμοδιότητέ τη λοιπόν η ορου οι Επιτροπή. Το πεδιο εφαρμογη τη βασικη νομοθετικη πραξη αυτο δεν επιτρεπεται εδω ξεπερνα τι αρμοδιοτητε τη λοιπον η ευρωπαικη επιτροπη το τελικό κείμενο και την προηγούμενη εβδομάδα, ε, να προσαρμοστεί μάλλον το κείμενο είχαμε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα, χρειάζεται να γίνει αυτό. Και επίση τα κείμενα θα πρέπει να είναι συμβατά και με την τελική συμφωνία που επετεύχθη. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο ζήτημα των 8 τζουλ. Επίσης, τις προάλλες στο, στην Ολλανδική τηλεόραση, στο News World, έγινε μια συζήτηση για τα μικρά και πολύ μικρά drone, τα οποία δεν μπορεί κανείς να σταματήσει δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά προστατευτικοί, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν ε, ε, να μην υπάρχει έλλειψη συνοχής στην νομοθεσία για τα τρόουν. Εγώ παίρνω πολύ στα σοβαρά τις διάφορες ανησυχίες που εξέφρασε ο κύριος Μαρινέσκου παρά από αυτά που μας λέει ο κύριος... Συγγνώμη, κυρία Φώστερ. Κύριε Κορνέλης, ε, θέλετε το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θέσαμε και σε αυτές που δεν θέσαμε. Στα Ολλανδικά όχι μάλλον, αλλά παρόλα αυτά τα, γνωρίζω να τα καταλαβαίνω. Θα ξεκινήσω... Ναι, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι βεβαίως μπορώ να σας στείλω την παρουσίαση. Επίσης, το non-paper μπορείτε να διαβάσετε ε, γιατί δίνει και κάποιες πληροφορίες επιπλέον, υποβάθρου, που δεν τις βρίσκει κανείς συχνά σε ένα νομικό κείμενο. Αυτή η πράξη κατ' εξουσιοδότηση δεν, κατα... δεν ε, συμπεριλαμβάνει προϋποθέσεις πιστοποίησης για όλες τις κατηγορίες. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι θα υπάρξουν άλλες νομοθετικές, αντίστοιχες μάλλον πράξεις, για τις υπόλοιπες ε, κατηγορίες drone, οι οποίες ε, είναι πιο περίπλοκα μηχανήματα, χρησιμοποιούνται σε πιο περίπλοκες συνθήκες και γι' αυτόν τον λόγο η ΆΣΑ χρειάζεται περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να ε, εξετάσει τους κανόνες. Όμως θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν επιτρέπεται η χρήση τέτοιων drone πριν να υιοθετηθούν οι σχετικοί κανόνες και πριν να υπάρξουν σχετικές πιστοποίηση. Τώρα, ναι, στην ανοιχτή κατηγορία συμπεριλαμβάνουμε ντρόουν μέχρι 25 κιλά, ωστόσο μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και περιορισμοί στη χρήση που μπορεί να γίνεται εάν θέλει κανεί να αναφερθεί σε ανοιχτή κατηγορία. Κατά βάση αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αυτό είναι η πεμπτουσία της προσέγγισης της βασιζόμενης στην αξιολόγηση κινδύνου, την οποία υιοθετήσαμε και, και εμείς και η Άσα. Το οποίο σημαίνει τι, ότι έχουμε έχουν ξεχωριστές νομοθετικές ρυθμίσεις όταν εμπλέκονται άνθρωποι και άρα μπορεί να κινδυνεύσουν άνθρωποι οι περιουσίες από ότι όταν δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για να μιλούμε για ανοιχτή κατηγορία δεν υπερίπταται ανθρώπων των drone. Εάν κάποιο θέλει να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο drone και ε, να το πετάξει πάνω από ανθρώπους θα χρειάζεται να λάβει ένα πιστοποιητικό. Τους σχετικούς κανόνες δεν τους έχουμε ακόμα. Αλλά ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτή η επικίνδυνη χρήση drone δεν επιτρέπεται. Εκτός βέβαια αν κανείς παραβιάσει τον νόμο. Τώρα, ε, ε, γι' αυτό που είπα για το να σεβαστούμε τη συμφωνία σε σχέση με τι ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι τη σεβαστήκαμε, αλλά βεβαίω μπορούμε να το συζητήσουμε και διμερώς. Να μου πείτε ακριβώς ποιες είναι οι διατάξεις που είτε εσείς είτε ο κύριος Μαρινέσκου πιστεύετε ότι δεν έχουν ενταχθεί στο σωστό νομοθετικό κείμενο. Ε, εγώ είμαι πεπισμένος ότι τα κάναμε σωστά, αλλά να το συζητήσουμε αν θέλετε. Για το ζήτημα των 8 τζάουλ. Ε, δηλαδή το να υπάρχει αυτό ως κριτήριο για την καταχώρηση. Ο κανονισμός της ΕΑΣΑ ανέφερε μια σειρά κριτηρίων. Τα 8 τζουλ είναι ένα από αυτά. 8 τζουλ ε, αντιστοιχεί περίπου σε 900 γραμμάρια, περίπου. Ε, αυτό που κάνουμε εδώ είναι να ακολουθήσουμε μια πιο επιφυλακτική, μια πιο προστατευτική προσέγγιση και να χαμηλώσουμε το όριο. Γιατί, γιατί υπάρχουν και επιπλέον κριτήρια στον ε, κανονισμό που έχουν σχέση με την ασφάλεια. Γιατί μας λένε ότι ακόμα και τα μικρά drone μπορούν να τύχουν, να χρησιμοποιηθούν για επικίνδυνους σκοπούς. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ζητούμε να καταχωρούνται, να καταγράφονται μάλλον ε, περισσότερα drone από ότι θα καταγράφονταν ένα απλώ αναφερόμενο σε 8 Joule. Και επίση προσθέτουμε και το εξή, θα πρέπει να καταγράφεται ένα ντρόν οποτεδήποτε έχει κάποιον αισθητήρα ή κάποιον καταγραφέα, γιατί αυτό δημιουργεί ανησυχίε για την ιδιωτικότητα. Τα κάνουμε όλα αυτά, κάνουμε όλε αυτέ τι προτάσει επειδή βασιζόμαστε στην αρχή τη προφύλαξη. Νομίζω απάντησα στα πιο σημαντικά από τα ερωτήματα που μου θέσατε. Ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε κύριε Κορνέλη. Το επαναλαμβάνω, δεν γίνεται να ξεκινήσουν να κυκλοφορούν 25 κιλών ντρόουν στον αέρα χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούνται ήδη τέτοια drone και μας λέτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να, περάσει, για να ελέγξει κανείς ένα χωράφι, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι και πρέπει να φροντίσουμε να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Και ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι ο κανονισμός είναι σε ισχύ. Έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πράξη λοιπόν κατά εξουσιοδότηση θα πρέπει να συμφωνεί με αυτό. Αυτό το έγγραφο απαιτεί τόσο πράξη καταξιοδότηση όσο και εκτελεστικές πράξεις. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Να σας πω επίσης ότι υπέβαλα επίσημη ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μου απαντήσει σχετικά με την συμμόρφωση ε, πράξεων καταξιοδότηση, εκτελεστικών πράξεων και βασικού κανονισμού. Και έλαβα μία απάντηση η οποία νομίζω πως ε, δεν με ικανοποίησε και χρειάζεται έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν θα ζητήσω, να γίνει έλεγχος. Και σίγουρα Μπορούμε μαζί με τον κύριο Κορνέλης να το δούμε, όμως οι διατάξεις βρίσκονται μέσα ε, στον ε, κανονισμό και δεν, υπάρχει κα... και δεν υπάρχει καμία διάταξη σχετικά με αυτές τις πράξεις καταξιοδότηση για την πιστοποίηση. Τώρα μας ε, λέτε για δευτερογενή νομοθεσία. Υπάρχει, προβλέπεται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανόνα ότι υπηρεσίες που θα παρέχονται από drones θα πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την πιστοποίηση επανδρομένων αεροσκαφών. Αυτό είναι στον εκτελεστικό ε, κανονισμό και στο non-paper αναφέρεται ότι αυτοί οι κανονισμοί θα προσαρμοστούν για να εφαρμοστούν στην περίπτωση των drones. Αυτά λοιπόν ως προς τη δευτερογενή νομοθεσία. Και για τα 8 τζάουλ δεν υπάρχει καμία διάταξη. Αυτό είχε ως σκοπό να καλύψει drones ε, με υψηλής ταχύτητας μέχρι 250 γραμμάρια και, αλλά και drones χαμηλής ταχύτητας πιο βαριά, περισσότερα από 250 γραμμάρια. Γι' αυτό λοιπόν ήταν τόσο επίμαχο το σημείο αυτό στις διαπραγματεύσεις. Και θεωρώ πως χρειάζονται διευκρινήσεις περαιτέρω. Κύριε Μαρινέσκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να λάβει εγώ την Προεδρία για να ολοκληρώσουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να φύγετε. Όχι, όμως πριν ε, σας ε, αναφέρω τα συμπέρασματά μου. Τόσο εσείς όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα είναι να συναντηθείτε διμερώς για ορισμένες λεπτομέρειες, ιδιαίτερα από, ε, σε ό,τι αφορά τις πράξεις καταξιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις και μετά ο κύριος Μαρινέσκου θα μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της διμερούς αυτής συνάντησης. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ε, Τζάκι, σύντομα παρακαλώ. Και χω, χωρίς καμία καθυστέρηση. Ορισμένε φορέ ο πρόεδρο ε, μαντεύει τι θα πει κυρία Φώστερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο τη ημερησία διάταξη. Η κυρία Ροντρίγκε είναι εδώ. Καλώς ήρθατε. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το πρωτόκολλο ε, που τροποποιεί την Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές με την Κίνα έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο κανονισμού η κυρία Ροντρίγκε από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, θα μιλήσω πορτογαλικά, γι' αυτό να φορέσετε τα ακουστικά σας όσοι δεν γνωρίζετε τη γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εξ ονόματο ε, του συναδέλφου, ο οποίο ε, δυστυχώ λόγω ασθένεια δεν μπόρεσε να έρθει και θα διαβάσω λοιπόν την ε, δήλωσή του. Κύριε Πρόεδρε, η πρόταση που παρουσιάστηκε σήμερα δεν έχει αμφιλεγόμενα σημεία, ό,τι έχει αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλα θέματα ισχύει και στην περίπτωση ε, της συμφωνίας με την Κίνα. Θα χρειαστεί τροποποίηση έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρωτόκολλο λοιπόν προβλέπει την συμπερίληψη της Κροατίας χωρίς κάποια μεγάλη αλλαγή. Την 1 Μαρτίου, 2008 ετέθησε ισχύ η συμφωνία αυτή. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την εντολή της τροποποίησης και το 2014 ε, εστάλει από την Κομισιόν η συμφωνία αυτή, το πρωτόκολλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 είχαν ολοκληρωθεί εργασίε έτσι ώστε το Συμβούλιο να ε, κυρώσει το πρωτόκολλο αυτό φέτος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην κυρία Λουβατσιεύσκα, σκιώδη ηγητή εξ ονόματος του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Πράγματι δεν υπάρχει κάτι το αμφιλεγόμενο στο έγγραφο αυτό. Η Κροατία προσχώρησε το 2013, γι' αυτό λοιπόν και χρειάζεται τροποποίηση του πρωτοκόλλου. Οποιαδήποτε εθνική συμφωνία χρειάζεται τροποποίηση για να λάβει υπόψη ε, την προσχώρηση νέου κράτους μέλους. Αυτό δεν είναι τίποτα το πρωτόγνωρο, είναι μια τυπική διαδικασία και δεν υπάρχουν Επίμαχη σημεία. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως όλες οι ομάδες θα υπερψηφίσουν την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ράντος, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να δώσουμε την πλήρη στήριξή μας στη σύσταση αυτή, λογικότατη, δεν αλλάζει την ουσία τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, θα δώσουμε την πλήρη στήριξή μας στην ε, σύσταση αυτή. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγγνώμη αν προφέρω λάθος το όνομά σας, ελληνικό φαντάζομαι, κύριος Δημητριάδης. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εμείς ε, καλωσορίζουμε αυτή την ε, πρόταση, το σχέδιο σύστασης ε, και ελπίζουμε να εγκριθεί γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όπως και στην περίπτωση του, της διεύρυνσης του 2004 αλλά και στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας 2017 είναι πολύ σημαντικό να ε, παρασκευθούν τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να προσθεθεί και η Κροατία στην συμφωνία αυτή. Έχουν γίνει ετήσιες συναντήσεις για την ε, συμφωνία αυτή με τις θαλάσσιες μεταφορές με την Κίνα και είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί λοιπόν και η δημοκρατία της Κροατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σαφέστατος ήσασταν. Κύριε Ροντρίγκε, θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια αυτά. Ε, να πω ότι ε, μίλησα εξ ονόματος του συναδέλφου, οπότε τα σχόλια είναι δικά του και όχι δικά μου. Σας ευχαριστώ. 6 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, και κατόπιν αυτού ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο της ημερησία διάταξης. Βλέπετε πόσο καλοί είμαστε εμείς οι Ολλανδοί στο να κρατάμε τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της ε, δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταφορών και θα συνεχίσουμε σε δύο λεπτά και κλεισμένων των θυρών που και θα γίνει ενημέρωση για τα αποτελέσματα των διάφορων τριμερών διαλόγων. Οδικές υποδομές, κυρία Γιούτο, εδώ είστε. Μετά Μαρινέτσκου και Τελίτσκα για το συνδέοντα στην Ευρώπη. Κύριε Τελίτσκα, είστε εδώ πολύ ωραία. Κύριε